Πιλάρ δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω το χέρι σου, λέει η πρόεδρος. 5,98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5,99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 601 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 602 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 603 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 604 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 605 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 606 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 607 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 608 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 609 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 610 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 611 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 612 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 613 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 614 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 615 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 616 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 617 υπέρ 6-17-6-18 μαζι κατά αποχές εγκρίνονται. 619 κατά αποχές εγκρίνονται. 620 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 621 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 622 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 623 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 624 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 625 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 626 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 627 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 628 υπέρ κατά απορρίπτεται. 629 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 630 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 631 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 632 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 633 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 634 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 635 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 636 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 637 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 638 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 639 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 640 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 641 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 642 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 είναι τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 2 του συγκητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 στα δύο τμήματα. 102 είναι, 102. Εγώ είδα μόνο το 10, δεν είδα το 2.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 Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 και 12 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 και 117 και 118 μαζί, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121, 22, 23 μαζί, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ, 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 136 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία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 48 υπέρ 7 κατά μία αποχή συγχαρητήρια στον εισηγητή για τις διαπραγματεύσεις αρχίζει Μπράβο κυρία Πρόεδρε, μπράβο! Αρχίζει η ψηφοφορία. Πρέπει να ψηφίσετε για τις διαπραγματεύσεις. Είναι ανοιχτή ψηφοφορία. Γιατί λείπουν ακόμη ένα σωρό ψήφι. Κανένας δεν θέλει να ψηφίσει πια. Α, έρχονται, έρχονται ψήφοι. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. 50 υπέρ 1 κατά δύο αποχές Συγχαρητήρια. Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Μπράβο συνάδελφε Μπελέτ. Non puoi Ο κύριο Κράμερ, λοιπόν, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 3. Αφαιρέθηκα, λέει η πρόεδρο. Η τροπολογία 2 χωρίζεται σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Έλωσο ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 23 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 10 του προϋπολογισμού υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την τροπολογία 10. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 36 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 59. Αρχίζει η ψηφοφορία. Έχουμε έναν σοσιαλιστή περισεβούμενο. Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ 28 κατά απορρίπτεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 63 δεν είναι σαφές. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για την 20 ηλεκτρονικά, γιατί 70 απορρίφθηκε. Τροπολογία 20 λοιπόν. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 71 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Για το δεύτερο μέρος ηλεκτρονικά. 28-26 εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Εμένα μου φαίνεται να έχει απορριφθεί, αλλά στο ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 47 υπέρ 6 κατά, καμία αποχή. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Πέντε λεπτά διάλειμμα για να φύγουν όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα και μετά συνεχίζουμε. questo non funziona. Allora ricominciamo i lavori. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις εργασίες μας και το λόγο έχει ο συνάδελφος το Ζενόφσκι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε αυτή την πρόταση που επανειλημμένα την έχουμε συζητήσει. Είχαμε και την τελευταία φορά μια ακρόαση που έγινε και σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε 54 τροπολογίες που κατατέθηκαν και με τους σκιώδεις εισηγητές 37 συμβιβαστικές τροπολογίες καταφέραμε να εκπονήσουμε, να διατυπώσουμε. Κάποιες τροπολογίες είναι διατυπωτικής βελτίωσης ή αφορούν χτένισμα του κειμένου και υποστηρίζονται πολλές από αυτές από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Έχουμε λοιπόν εδώ τις προτεραιότητες που τονίζουμε Έχουμε συζητήσει λοιπόν αρκετά αυτό το θέμα κατά το παρελθόν. Πρόκειται για τους στόχους της ψηφιακής, του ψηφιακού θεματολόγιου της ψηφιακής ημερήσιας διάταξης. Μπορούμε να δεχθούμε αυτές τις προτάσεις. Είναι σημαντικό να καταφέρει να επιτύχει αυτούς τους στόχους η Ευρώπη ώστε να είναι παγκόσμια ανταγωνιστική και να μπορέσει να αντέξει τον ανταγωνισμό πρέπει το τεχνικό επίπεδο να παραμείνει στο ανώτατο επίπεδο και να μπορέσει να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να μεριμνήσουμε να παραμείνει η παραγωγή στην Ευρώπη με έδρα την Ευρώπη και ευρωπαϊκές βιομηχανίες με έδρα τις ευρωπαϊκές χώρες. Ζητούμε να υπάρχει πρόσβαση και σύνδεση ταχύτατα με το διαδίκτυο. Αυτό θα πρέπει για όλα τα νοικοκυριά να είναι εφικτό τουλάχιστον για ένα με πολύ μεγάλο αριθμό αυτών των οικοκυριών που θα μπορούν πρέπει να μπορούν να συνδεθούν με το διαδίκτυο. Να ανταποκριθούμε στις προτεραιότητες λοιπόν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τις διατυπώσεις στις οποίες καταλήξαμε, ώστε εκείνοι που επιθυμούν να μπορούν όλοι να έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια τέτοια πρόσβαση. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε για ελαστικότητα και πολυμορφία πολυσχηδή χαρακτήρα των σχεδίων και προγραμμάτων. Οι όροι και προϋποθέσεις διαφέρουν από κράτος σε κράτος. Πολλά κράτη-μέλη σήμερα έχουν καλά προετοιμαστεί και έχουν προετοιμάσει αυτά τα, αυτές τις υποδομές και τα πράγματα βαίνουν καλό. Σε, άλλα, σε άλλες χώρες ε, δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ. Πρέπει τεχνολογικά να είμαστε αμερόληπτοι και ουδέτεροι. Είναι σημαντικό να έχουμε την τεχνολογία και να διασφαλίσουμε και τα κονδύλια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τα βέλτιστα σχέδια και προγράμματα. Το τεχνολογικό επίπεδο πρέπει να αναβαθμιστεί και να καταφέρουμε εκεί όπου έχουμε τα καλύτερα, τα βέλτιστα αποτελέσματα να είναι ανωτά του επίπεδου. Είναι χρήσιμο, πιστεύω, να συζητήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα της ζήτησης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όχι μόνο οι σημερινές ανάγκες των καταναλωτών είναι ε, μια σημαντική υπόθεση, αλλά η ζήτηση διαμορφώνεται όλο και αλλάζει, ώστε στο μέλλον αυτά θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Δεν μπορούμε να μιλάμε και να αναφερόμαστε στη σημερινή, στα σημερινά επίπεδα ζήτησης, διότι οι εξελίξεις ακολουθούν ταχύτατους τους ρυθμούς και αυτό ισχύει και παγκόσμια. Αυτό που πριν από έξι μήνες ήταν επίκαιρο, τώρα μπορεί να θεωρείται ανεδαφικό και παροχημένο και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε και για το μέλλον για τις μελλοντικές πρόπτικες και έτσι θα πρέπει αυτή την τροχιά, αυτή την πορεία να προετοιμάσουμε και να είμαστε έτοιμοι. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέρφους, τον κύριο Χέκμακ, την κυρία Τροθμάν, την κυρία Άντερς Ντότερ επίσης. Οι συνάδελφοι με υποστήριξαν όσον αφορά το εγχείρημα αυτό και καταφέραμε πραγματικά διεξοδικά να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα χάρη στις δικές, τις δικές τους προτάσεις εμπλουτίστηκε και έγινε καλύτερο αυτό το έγγραφο. Προσπάθησα κάποιες τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες να τις συμπεριλάβω ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έγκριση με την ψηφοφορία. Η ψηφοφορία προς έγκριση προβλέπεται για την 5η Νοεμβρίου. Και στη συνέχεια τον Ιανουάριο πιθανότατα του 2013 θα καταλήξει το θέμα στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Οι σκιώδεις συζητητές έχουν το λόγο. Συνάδελφος Όκμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και πάλι και συγχαρητήρια στον κύριο Τοζανόφσκι του οποίου η έκθεση θεωρώ ότι τονίζει τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να εξειδικεύσουμε τους στόχους μας. Έχουμε συζητήσει ορισμένα από τα θέματα αυτά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχετικά με το ευρέω φάσμα του διαδίκτυο στην Επιτροπή μας. Αυτό που με ανησυχεί και νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει το βάθρο για την συζήτησή μας, τη βάση για τη συζήτησή μας, είναι το γεγονός ότι μεγάλα μέρη της πιο δυναμικής ανάπτυξης σχετικά με το διαδίκτυο και το ευρύ φάσμα δεν λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη. Η Νότια Κορέα, μια από τις μεγάλες αναφιόμενες ασιατικές οικονομίες είναι αυτή που ηγείται. Βέβαια βλέπουμε και ότι μετά από αυτήν έρχονται για παράδειγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ε, το Χονγκ η Ιαπωνία, η Ταϊβάν. Ίσως είναι σχετικά μικρά μέρη της οικονομίας, αλλά αποτελούν ωστόσο μια εξέλιξη που είναι, που αποτελεί σημαντική πρόκληση. Ενώ εμείς στην Ευρώπη κινδυνεύουμε να μην είμαστε διόλου το νούμερο ένα, ίσως ούτε και το νούμερο δύο, να είμαστε τρία ή τέσσερα. Από τη δική μου σκοπιά, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ δεν πρόκειται μόνο για την ε, χωρητικότητα του ευρωσφάσματος ή την ταχύτητα, αλλά για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Εδώ και λίγο σχετικά χρόνο είχαμε μεγάλη, τη μεγάλη ικανοποίηση να μπορούμε να στέλνουμε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, γράμματα δηλαδή, αν θέλετε να το πείτε έτσι, και ίσως θυμάστε ότι ε, το η οθόνη ήταν πράσινη και τα γράμματα κίτρινα. Τι ωραία που ήταν. Αλλά ήταν διαφορετική υπηρεσία από αυτήν στην οποία έχουμε συνηθίσει πλέον σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη χωρητικότητα, capacity, θα καλύπτεται όλο και γρηγορότερα από νέες υπηρεσίες, όπως είναι αυτές οι εφαρμογές, οι applications. Με εντυπωσιάζει το γεγονό ότι στην Ιαπωνία ε, κάνουν τώρα δοκιμές οπτικών καλωδίων πώς να σας το πω που ε, προωθούν 14 τρισεκατομμύρια bit το δευτερόλεπτο. Είναι ασύλληπτο το μέγεθος αυτό. Είναι, τι να σας πω, πάρα πάρα πολύ. 14 τρισεκατομμύρια είναι σαν 14 τεραμπάιτ που είναι χίλιες ώρες περισσότερο από ένα γίγαμπάιτ. Και δεν νομίζω βέβαια ότι αυτό θα είναι και το σύνηθες, αλλά δείχνει ότι πηγαίνουμε τα όρια της τεχνολογίας όλο και μακρύτερα. Και από την δική μου σκοπιά είναι σημαντικό όταν θα βάλουμε στόχους, όταν θα ορίσουμε στόχους για τις μελλοντικέ μας χωρητικότητες και στην Ευρώπη, θα πρέπει να σκεφτόμαστε με ορίζοντα το 2020 και όχι το 2012. Τα επιτεύγματα του 2012 θα είναι πλέον ιστορία το 2020. Είναι σαν να σας ζητήσω να κοιτάξετε πίσω τι γινόταν το 2004 και την ταχύτατη εξέλιξη που είδαμε στο μεταξύ. Πάλι όχι τόσο πολύ την ε, αύξηση της χωρητικότητας ως τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά τις υπηρεσίες που μπορούμε να βασίσουμε σε αυτά. Και αυτά θα αποδώσουν μετά την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα στις οικονομίες μας. Πρόκειται για έναν από τους κρισιμότερους τομείς για την αγωνιστικότητα της Ευρώπης και για την ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής μας οικονομίας και της οικονομίας υπηρεσιών, αλλά που θα καταστήσει επίσης δυνατή τους ε, telecom operators στην ε, Ευρώπη και όλες τις άλλες σχετικές επιχειρήσεις να αναλάβουν ηγετικό ρόλο. Σε ό,τι αφορά τώρα τους στόχους, νομίζω ότι οι συμβασμοί που ε, περιέγραψε ο κ. Στανδρόφσκι είναι καλοί. Δεν θέλω όμως να αποδυναμωθούν. Και θα σας πω για, ποιο, για ποιους τρεις λόγους. Πρώτος, οι στόχοι μας συνδέονται τώρα πλέον με κριτήρια. Δηλαδή οι στόχοι που καθορίζουμε θα έχουν κάποιες επιπτώσεις στην πραγματικότητα. Χαμηλή στόχη, χαμηλές εξελίξεις. Υψηλή στόχη, υψηλότερη, ταχύτερη εξέλιξη. Όπου θα, θα, θα συνδέσουμε μάλλον ε, τις δαπάνες με τα κριτήρια. Εγώ πιστεύω ότι η δική μας ευθύνη είναι να διασφαλίσουμε ότι οι μεγάλες πόλεις μας, τα πανεπιστήμια μας, οι πανεπιστημιακές μας πόλεις θα έχουν την υψηλότερη χωρητικότητα στον κόσμο, γιατί αυτό αποτελεί προπόθεση για να παίξουμε ηγετικό ρόλο. Αν δεν το θέλουμε αυτό, βέβαια μπορούμε να βάλουμε χαμηλότερου στόχου. Αλλά νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε επ' αυτού. Το ίδιο πιστεύω, και αυτό είναι ο δεύτερος λόγος, ότι όταν αν καθορίσουμε τώρα τους στόχους, στην ουσία καθορίζουμε και τις διαθρώσεις του 2020, γιατί η επενδύσεις που θα γίνουν σήμερα θα είναι δύσκολο να αντικατασταθούν σε 2-3 χρόνια στο μέλλον. Αν λοιπόν είναι πολύ χαμηλά τα κριτήρια και οι στόχοι μας σήμερα, τότε αυτοπεριοριζόμαστε σε μια, μια ανταγωνιστική υποδομή για το ευρύ φάσμα και το διαδίκτυο. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε ήδη σε διάφορα σημεία της Ευρώπης όπου έγιναν επενδύσεις στο ευρύ φάσμα, όμως ιστό συγγνώμη, στόχοι ήταν υπερβολικά χαμηλοί. Και δεν μιλώ για περιοχές της Υπέθρου. μιλώ για περιοχές πυκνοκατοικημένες και με μεγάλη οικονομική ε, ανάπτυξη. Όμως ήταν πολύ χαμηλοί οι στόχοι και τώρα έχουν αυτοπεριοριστεί μέσα σε περιορισμένες χωρητικότητες που δεν τους προσφέρουν επαρκείς ευκαιρίες. Και ο τρίτος λόγος που βρίσκω ότι είναι σημαντικός, εάν όντω είμαστε σοβαρή σε ό,τι αφορά την υπέρβαση του ψηφιακού χάσματος είναι ότι και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι 2015, 2017, 2020 και οι περιοχές της Υπέθρου πρέπει να μπορέσουν να παρακολουθήσουν. Δηλαδή χρειαζόμαστε εκεί την ευκαμψία που ανέφερε ο εισηγητής χωρίς ταυτόχρονα να απόσχουμε από τους στόχους. 100 GB για τις πυκνοκατοικημένε περιοχέ και 100 GB για τις περιοχέ υπαίθρου που αλλιώ θα παραμείνουν ε, περιοχέ απομονωμένες όπως είναι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Κατρίν Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία. Πρόκειται για μία τριπλή πρόκληση. Πρόκειται για την κάλυψη του ευρωπαϊκού χώρου από αυτήν την υπηρεσία, όπως επίσης και να συμβάλλουμε στην ανάκαμψη, στην οικονομική ανάκαμψη υπέρ των συμπολιτών μας στην Ευρώπη. Εμείς ε, με αυτή την έκθεση θα πρέπει να ε, δούμε την αποτελεσματικότητα της έκθεσης, διότι άμα η έκθεση δεν είναι αποτελεσματική, είναι σαν να δίνουμε, ε, σαν κάνουμε τρύπες στο νερό. Διότι αυτό το οποίο μας χρειάζεται είναι και η ανταγωνιστικότητα. Έχουμε μια άλλη πρόκληση να μην μειωθεί το ποσό το οποίο αφιερώνεται στις τηλεπικοινωνίες και στις νέες τεχνολογίες. Θα ήθελα να, να αναφέρω τα σημεία εκείνα με τα οποία διαφωνούμε, ποια συνεχίζουμε να συζητάμε και μερικά στοιχεία. Λοιπόν, εμείς συμφωνούμε σε τρία πράγματα διαφορετικού μεγέθους πρόταση για τους, την ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα πλαισιώνει την Κομισιόν. Σήμερα έχουμε συνένεση και για το πεδίο αρμοδιοτήτων αλλά και για τους τομείς που θα καλύπτονται από αυτούς τους εμπειρογνώμονες. Μετά σε συνέργεια με άλλους τομείς, ενέργεια και μεταφορές που πρέπει να ευνοήσουμε. Προσέχοντας όμως να μην επικαλύψουν τον τομέα μας. Επίσης, συμφωνούμε να συμπεριληφθούν στο ΣΕΦ οι τοπικές αρχές. Για το θέμα των στόχων. Εγώ καταλαβαίνω την βούληση του κυρίου Χόχμαρκ και του εισηγητή για την φιλοδοξία που έχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν η Κομισιόν μας λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να προσεγγίσουμε τους στόχους της ατζέντα. Αν εμείς όμως επιμείνουμε στο ψηφιακό, τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να περιορίσουμε τους άλλους τομείς και άμα εμείς υπερχρηματοδοτήσουμε τότε δεν, είναι, δεν βλέπουμε δυνατότητες έλξης του ιδιωτικού τομέα και φυσικά δεν θα βοηθήσουμε αυτούς που σήμερα δεν μπορούν να αναπτύξουν ένα πραγματικό δίκτυο με χαμηλής ταχύτητας. Παρακαλώ λοιπόν να μην αγνοήσουμε τις τοπικές και κοινωνικές ανάγκες της Ένωσης, διότι τότε θα έχουμε χάσει την αποτελεσματικότητά μας. Επίσης, στις χώρες εκείνες όπου αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει, τουλάχιστον να λειτουργήσει διασύνδεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τα σχέδια εκείνα, να προθίσουμε τα σχέδια εκείνα τα οποία ξεπερνούν το 1 GB ε, ανά δευτερόλεπτο. Επίσης, πρέπει να γίνει μία ανάλυση αγοράς πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα και συμφωνούμε σε αυτό. Δεν θα πάμε να επενδύσουμε εμείς εκεί όπου οι ιδιώτες μπορούν να επενδύσουν. Αλλά και αυτή η φάση διερεύνησης δεν μπορεί να κρατήσει επάπειρον. Και δεν μπορούμε εμείς ε, να αργήσουμε να μείνουμε καθυστερημένοι εκεί όπου δεν παρεμβαίνουν τα ιδιωτικά κεφάλαια. Τώρα για το θέμα των τελεκόμ των τηλεπικοινωνιακών εταιριών και των υπηρεσιών. Αυτό πρέπει να ενταχθεί μέσα στη λογική της ανάκαμψης και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν ποιες προσπάθειες εμείς απαιτούμε και πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά. Επίσης έχουμε έναν άλλο στόχο που θα ήθελα να σας ε, θυμίσω συμπερασματικά είναι να μπορέσουμε να καλυφθούμε εγκάρσια. Δεν μπορούμε εμείς ε, να αγνοήσουμε τις guidelines άμα δεν έχουμε ορίσει τους ε, στόχους και τις εφαρμοστικές λεπτομέρειες και δεν, στεκόμαστε, και δεν έχουμε καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές. Και αυτό για να μην βρεθούμε σε αντίφαση στο τέλος για τις λεπτομέρειες, δηλαδή για το ρόλο που θα πρέπει να παίξει η ΕΤΕ και τα κράτη-μέλη, φαίνεται να, κάτι να διαγράφεται στο Συμβούλιο. Εμείς θα πρέπει να διαμορφώσουμε στο Κοινοβούλιο μια κοινή θεωρία μεταξύ των διαφόρων επιτροπών και των διαφόρων εισηγητών πριν από τον Τρίλογο, διότι αν εμείς καταφέρουμε να συγκλίνουμε μεν, δεν θα έχουμε τελειώσει τη δουλειά μας στην εποχή αν δεν καταφέρουμε να συγκλίνουμε δεν θα έχουμε τελειώσει τη δουλειά μας για να προετοιμαστούμε στις συναντήσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ο Γιούργεν Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου προηγουμένως, επιθυμώ και εγώ να δηλώσω την ε, συνένεσή μου για τις τροπολογίες συμβιβασμού. Νομίζω κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, έστω και αν υπάρχουν ορισμένα ζητήματα επί των οποίων διατηρώ επιφυλάξεις. Και τονίζω επίσης ε, ότι έχουμε επιφυλάξεις ως ομάδα σε ό,τι αφορά την καταβολή ενισχύσεων. Θα έπρεπε τα συνηθισμένα χρηματοδοτικά μέσα να αρκούν. Επίσης είναι σημαντικό για μένα η αναμενόμενη ζήτηση να λαμβάνεται υπόψη όταν απολαμβάνονται αποφάσεις για τα έργα αυτά. Είπα και στην πρώτη συζήτηση ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι γενικά σε τμήματα της υπαίθρου έχουμε μείωση του πληθυσμού. Άρα πρέπει οι μεγάλες αυτές ύψους εκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις να γίνουν εκεί όπου είναι δικαιολογημένο. συνειδητά δεν παραμελούμε την Ήπεθρο, διότι οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις συχνά εγκαθίστανται στην περιφέρεια και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να διαθέτουν καλή ε, πρόσβαση σε ευρυφασματικό διαδίκτυο για να μπορέσουν να προωθήσουν ε, την παραγωγή τους. Είπαμε, είπαν άλλοι προηγουμένως ότι πρέπει να έχουμε φιλόδοξους στόχους οι οποίοι να καλύπτουν και το 2020 και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και τότε. Από την άλλη μεριά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Εφόσον όμως ε, βάλουμε οι πολύ ψηλές απαιτήσει και μετά δεν προκύψει η ιδιωτική επένδυση, διότι δεν υπάρχουν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι, τότε πάλι και αυτό θα είναι λάθος. Τότε δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή ναι μεν φιλόδοξη στόχη, αλλά παρόλα αυτά ρεαλιστική. Και να μην προσανατολιστούμε σε στόχους που ίσως είναι δυνατόν να επιτευθούν σε μεγάλα αστικά κέντρα όπου είναι πολύ πυκνά τα δίκτυα και επομένως πολύ πυκνά τα δίκτυα και της ζήτηση, αλλά να γίνει κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των αστικών κέντρων και των χώρων της περιφέρειας. Σημαντικό επίσης είναι να διαφυλάξουμε και την τεχνολογική ουδετερότητα. Έχουμε σχετικό ορισμό της ανοιχτής πρόσβασης. Σε αυτόν τον ορισμό πρέπει να βασιστούμε και να μην δημιουργήσουμε νέους ορισμούς. Τέλος, για τηλεπικοινωνία και την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Στις συζητήσεις περί προϋπολογισμού, οι χώρες μέλη προτείνουν και άλλες περικόπες και φαίνεται το τμήμα των τηλεπικοινωνιών να είναι το πρώτο του θύμα. Εγώ υπογραμμίζω τα όσα, όσα είπαν οι προαναλύσαντες ότι για την Ευρώπη είναι σημαντικό να παίξει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό. Και εάν θέλουμε η Ευρώπη να έχει κάποιο νόημα, θα πρέπει να υπάρχει και κάποια αντιστάθμιση μεταξύ χωρών μελών, ισχυρών χωρών μελών και λιγότερο ισχυρών, που ειδικά αυτές έχουν ανάγκη από την στήριξη των ευρωπαϊκών μηχανισμών. Και γι' αυτό πρέπει όλοι να το ξανασκεφτούν αυτό όσοι θεωρούν ότι πρέπει να περικόψουν τον προπολογισμό, να ξανασκεφτούν δηλαδή αν αυτό όντω είναι προ το συμφέρον τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και εγώ επίσης να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή τον κύριο Τοσνόσκη για τη δουλειά του για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Οι συμβαστικές τροπολογίες συζητήθηκαν μεταξύ των συντονιστών και δεν είναι μικρό το επίτευγμα. Έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση που αντανακλά τις περισσότερες παρατηρήσεις που έγιναν από εμάς σε σχέση με αυτά τα θέματα. Δυστυχώς και αναφέρθηκε αυτό το δίκτυο των τηλεπικοινωνιών, το Europe Connecting Facility, βρίσκεται υπό την πίεση των διαπραγματεύσεων, των διαβουλεύσεων για τα κονδύλια του προπολογισμού. Είναι σαφέ ότι από πλευρά δομή και για τι ηλεκτρονικέ υπηρεσίε ε, για την Ευρώπη και οι ευκαιρίε που χρειάζονται είναι πολύ σημαντική υπόθεση να ασκήσετε πίεση στα κράτη-μέλη γι' αυτό για να διαφυλαχθεί, να διασφαλιστεί αυτό το πρόγραμμα. Υποστηρίζω τους φιλόδοξους στόχους που προτείνονται από τον κύριο Χέρτμαρκ. Είναι καλό να είμαστε φιλόδοξοι και να υπάρχει αυτή η φιλοδοξία για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν από τον κύριο Χέρτμαρκ και όλους τους άλλους που τοποθετήθηκαν σε αυτά τα θέματα σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και οι ευρύτερε προτάσεις για τη διασύνδεση των χωρών της Ευρώπης και επίσης οι συμβαστικές τροπολογίες αφήνουν χώρο ε, λιγμών και δράσεις ε, για τους Δήμους, κοινότητες, ε, την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να μπορέσουν να δράσουν. Οι, οι δυνατότητες αυτές είναι ένα, πολύ καλό στοιχείο για να μπορέσει να αναπτυχθεί η Ευρώπη. Επίσης όσον αφορά τις υποδομές το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την παροχή υπηρεσιών Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Χονγκ για παράδειγμα είδαμε ότι μεγάλα δίκτυα υψηλής ταχύτητας και η κάλυψη αυτών σε αυτές τις χώρες είναι πολύ υψηλή και πολύ μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να διασφαλιστεί από πλευρά υπηρεσιών η δυνατότητα ε, ανοίγματο ε, για τον ανταγωνισμό στην αγορά, σε, ιδιαίτερα στις ε, οψιμότερες, στις ιστερότερες φάσεις. Θα ήθελα να διαφοροποιηθούμε λοιπόν επ' αυτών στις συμβαστικές τροπολογίες. Υποστηρίζουμε απόλυτα τις, ομάδες, τις προτάσεις της ομάδας υψηλών πραγματογνωμόνων, υψηλών αξιωματούχων. Πρέπει οι ε, πάροχοι και οι εμπλεκόμενοι να καλύπτονται και είναι καλό το ότι υπάρχουν σύμβαση προτάσεις τροπολογιών επ' αυτών. Στις υπηρεσίες και αυτό δεν συζητήθηκε στις διαπραγματεύσεις των συντονιστών αρχικά πρότεινε Πολλά πράγματα για την προστασία παιδιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλουν να καλυφθούν με τον προϋπολογισμό για τις υπηρεσίες αυτές. Θέλω να διαγράψουμε τα περισσότερα από αυτά εκτός από την υπεύθυνη χρήση σε σχέση με τη διασύνδεση. Αυτό εν μέρη, επειδή δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ο πιο ενδεδειγμένο προπολογισμό για τέτοιου είδου υπηρεσίε. Ζητήθηκε επίση και το Child Online σε σχέση με αυτό το εγχείρημα. Πολλά από τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν από αυτέ τι προποθετημένες υπηρεσίε, Δεν είναι τα προβλήματα εκείνα τα οποία θα αντιμετώπιζαν χαρακτηριστικά τα παιδιά χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Πρέπει καλύτερα να δούμε τις αξιολογήσεις, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα των παιδιών στο διαδίκτυο. Προτού δώσουμε και ένα σχετικά ευρύ μεγάλο προϋπολογισμό για να επιληθούν τέτοιου είδους προβλήματα. Υπάρχουν περισσότερα, περισσότερα χρήσιμα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με τέτοια κονδύλια, ιδιαίτερα τώρα και ιδιαίτερα αν υπάρξουν και περικοπές για τον προϋπολογισμό ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ. Grazie, Η e Pilar del οπότε αρχίζουν οι τοποθετήσει. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Τωσανόφσκι και εγώ για τη δουλειά που έκανε αυτός και οι σκιώδεις εισηγητές που και αυτούς ευχαριστώ που έχουν η μεγάλη σπουδαιότητα αυτό το έργο. Εγώ μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν που με αυτά ουσιαστικά συμφωνώ με μεγάλα τμήματα των παρατηρήσεων που έγιναν θα ήθελα λοιπόν να πω ότι μου φαίνεται ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα ωφέλη από μια τέτοια δράση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προάγει την διασύνδεση όσον αφορά δίκτυα και τα δίκτυα στην Ευρώπη μεταφορών, επικοινωνιών και άλλων και τώρα εδώ έχουμε τις τηλεπικοινωνίες είναι έχει τεράστια σημασία. Ιδιαίτερα στον τομέα όπου κινούμαστε τώρα εδώ. Κανείς δεν έχει καμιά αμφιβολία. Έχουμε προσωπικά βιώματα ότι η διακίνηση δεδομένων μέσω αυτών των δικτύων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα μέχρι το ίστατο σημείο ότι και σύμφωνα με πολύ διαφορετικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί με χρονορίζοντα το 2017-2018 δίνουν μια εκθετική ανάπτυξη ιδιαίτερη σπουδαιότητα, Οι ανάγκες των ε, συχνοτήτων, του εύρου συχνοτήτων, της ταχείας μεταβίβασης, διάδοσης δεδομένων όσον αφορά ε, τη διαβίβαση και μεταβίβαση αυτών των στοιχείων, των δεδομένων. Όλοι τα γνωρίζουμε αυτά, δεν χρειάζεται να επιμείνουμε περισσότερο από αυτόν. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα άλλο σημαντικό θέμα που πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ. Και αυτό είναι το ότι όχι μόνο θα πρέπει να ανοίξει η πόρτα για την χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων, για την ανάκτη, α, χρήση τέτοιων ε, ευρυζωνικών δικτύων ταχείας διαβίβασης στοιχείων και δεδομένων, αλλά επίσης, και αυτό είναι σημαντικό διότι ανοίγει ένα περιθώριο ελιγμών και ε, κινήσεων για τις διάφορε υπηρεσίε, Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνουμε και να εμείνουμε ιδιαίτερα στην δυνατότητα αυτά τα προγράμματα και σχέδια να συνδέονται με τις υπηρεσίες, με την παροχή υπηρεσιών. Η παροχή ε, ψηφιακών υπηρεσιών όσον αφορά την δημόσια διακυβέρνηση και στις ανάγκες μεθοριακών περιοχών είναι θεμελιώδους σημασίας. Θεμελιώδους σημασίας και επίσης τα σχέδια, τα προγράμματα μπορούν να λαμβάνουν αυτά όλα υπόψη. Έχει περιγράψει και κινηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέπει να κλείσουμε τις πόρτες και δυνατότητες ε, για κάποιες δράσεις. Υπάρχει ένα στοιχείο που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Η δρομολόγηση μιας ψηφιακής υπηρεσίας δημιουργεί άμεσα, άλλη άμεσα, ένα δυναμισμό, μια δυναμική, μια προώθηση που προκαλείται και νέε ανάγκες που αναφύονται και για τους καταναλωτές εξίσου όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών και τα λοιπά και όλα αυτά. Και έτσι υπάρχει και μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ανάγκη ως κύματα που εκφράζονται και αναφύονται. Έχουν τεράστιες επιπτώσεις όλα αυτά, όχι μόνο σε συγκεκριμένη υπηρεσία, σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία, αλλά άμεσα ξεκινά εδώ μια αλυσίδα αντιδράσεων, δημιουργείται μια νέα κατάσταση στο σύνολο του τομέα αυτού και στους συναφείς ε, όμορους ε, τομείς. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σε όλα αυτά. Τους δίνουμε σημασία όταν έχουμε το θέμα της δρομολόγησης ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά πρέπει να εμείνουμε σε αυτή την πτυχή. Τέλος, επιτρέψτε μου να τονίσω, να υπογραμμίσω ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλα αυτά. Θέλω να απευθύνω μια έκκληση σε όλους τους συναδέλφους μου <clears throat> ώστε να αποφύγουμε το, τα κονδύλια που προβλέπονται ε, ένα δις 200 εκατομμύρια ευρώ αν δεν κάνω λάθος <clears throat> για αυτό το κομμάτι των δικτύων και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο όλων των δράσεων που θα πρέπει να αναλυφθούν για την διασύνδεση της Ευρώπης, Connecting Europe Facilities, να μην μειωθούν όλα αυτά, να μην περικοπούν. Να μην υπάρξει συρρήκνωση, να μην πάνε σε άλλους τομείς όπως για παράδειγμα π.χ. στις μεταφορές και τα δίκτυα μεταφορών. Διότι διαφορετικά στο τέλος τι θα γίνει. Είναι προφανέ ότι πάντα υπάρχουν ανάγκε στον τομέα των μεταφορών, σίγουρα, αλλά δεν μπορούν όλα αυτά να καλύπτονται ει βάρο αυτών που προβλέπονται σε σχέση με τι προτάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικά μα δίκτυα, να μην μειωθούν αυτά τα κονδύλια για τι χρήσει που προβλέπουμε εμεί. και σε επαφή με τις, ε, την ίδια την κυβέρνηση ε, τη χώρα μα και απευθύνω έκκληση στα μέλη τη κοινοβουλευτική μα επιτροπή, να έρθουν σε επαφή με τι δικέ του κυβερνήσει, να μην υπάρξει όχι μόνο συρρήκνωση του συνόλου των κονδυλίων του Ταμείου και θα πρέπει στο Συμβούλιο να επαναδιαπραγματευτούμε όλα αυτά. Το, στο Ταμείο, στα κονδύλια, να είναι σεβαστές οι προτάσεις τη Επιτροπής για κάθε τομέα ξεχωριστά. Όλα αυτά είναι τα πιο σημαντικά νομίζω. Αυτά είναι, αυτή είναι η πιο σημαντική διαφοροποίηση και παρατήρηση. Να μην υπάρξει αυτή η σβάρος εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών στον τομέα των διαδικτύων. Ευχαριστώ. Sì, eh, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς έχουμε ένα θέμα που αφορά στα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνίας και εντάσσεται αυτό μέσα, στην ε, συνολική, μέσα στα πλαίσια των μεταφορών Ενέργεια στήλη επικοινωνιών. Είναι ένα τρίπτυχο. Εδώ έχουμε 9,2 δις ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι απέχουμε παρασάγκας από τις ανάγκες της Υπήρου μας. Διότι εμείς εδώ εκτιμούμε 100 με 150 δις ευρώ τις πραγματικές ανάγκες. Σίγουρα εμείς ε, πρέπει να το προωθήσουμε αυτό το ντοσιέ γιατί το έχουμε στο τραπέζι. Αλλά θα πρέπει πραγματικά να αναρωτηθούμε αν μέσα στα πλαίσια αυτού του μεγάλου σχεδίου υποδομών που μαζεύει πολιτική συνένεση Μήπως ε, θα μπορούσε στα πλαίσια του 2020 να έχει ποσά τα οποία ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της Υπήρου μας. Διότι δεν διέπεται ε, αυτό το σχέδιο από τη λογική της αγοράς και θα ήθελα να συμφωνήσουμε για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η αγορά δεν καλύπτει τις ανάγκες, τότε το δημόσιο θα πρέπει να παρέμβει για να διασφαλίσει τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε αυτά τα δίκτυα για τους πολίτες, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και εμείς έχουμε νομική βάση σχετικά με την επικρίτηση τις περιφέρειες εκείνες οι οποίες ε, έχουν πρόβλημα απόστασης, κυρίως δε τα, τα βουνά και τα νησιά και πρέπει να επιδείξουμε ευρωπαϊκή ελληνική σχετικά για την χρηματοδότηση, διότι πάντοτε υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης. Εγώ θεωρώ ότι δεν περνάμε ε, χρόνο όσον ε, ε, εξέτασης και αναζήτησης των θεμάτων χρηματοδότησης. Βρισκόμαστε στον 20ο αιώνα, εδώ είχαμε <clears throat> τον 20ο αιώνα, είχαμε τεράστιες τεχνολογικές πρόοδους από την ατμομηχανή μέχρι το πλυντήριο ρούχων. <coughs> Και στον 21ο αιώνα θα έχουμε πρόοδους. Ε, δεν μπορούμε να μείνουμε στο περιθώριο και να μην καλύπτουμε ορισμένα εδάφη. Και για παράδειγμα η χώρα μου φώτισε την Ήπεθρο δηλαδή έδωσε, έδωσε ηλεκτρισμό ε, στην Ήπεθρο με ένα μικρό ποσό επιπλέον στο τιμολόγιο της, ε, ε, του, ηλεκτρισμού. Μήπως αντίστοιχα και στην, σε τηλεπικοινωνίες, μήπως θα έπρεπε να βρούμε κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε για φόρο. Μιλάμε απλώς για αλληλεγγύη όπου ο πολίτης καταβάλει κάτι εγώ είμαι μεγάλη μειονότητα ε, στην ομάδα μου, γιατί κάθε φορά που μιλάμε για φόρους βγάζουν σπηριά. Αλλά αν εμείς θέλουμε να, ε, να, να ανταποκριθούμε στις ελπίδες που τρέφουν οι λαοί, θα πρέπει να βρούμε και τους σωστούς μηχανισμούς μεταξύ αγοράς, ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και χρηματοδότησης. Ευχαριστώ κύριε Οντίκε για τις προτάσεις σας. Το λόγο στην Κομισιόν να καλωσορίσω και τον νέο Διευθυντή των Τηλεπικοινωνιών, τον ε, δόκτορα Ρομπέρτο Βιόλα, ο οποίος ε, παίρνει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ στα αγγλικά. Κυρία Πρόεδρε, τιμή μου να βρίσκομαι εδώ μπροστά σας έχω ξαναέλθει στο Κοινοβούλιο και προηγούμενα υπό την παλαιά μου ιδιότητα που ήμουν πρόεδρος της ομάδας των ρυθμιστών, των ρυθμιστικών αρχών δηλαδή, για πρώτη φορά τώρα βεβαίως ως αξιωματούχος της Επιτροπής. Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που μου δίνεται αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ τον εισηγητή καθώς και τους σιώδης εισηγητές και τους άλλους ευρωβουλευτές και για την δουλειά που έχουν κάνει αλλά και για τη σημερινή συζήτηση. Σήμερα εμείς ακούμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ακούμε τη σημαντική αυτή συζήτηση αφού βεβαίως έχουμε διαβάσει πρώτα την έκθεση και τη συνέχεια που της έχει δοθεί. Είναι μεγάλη σημασία του προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το CFICT είναι χρήματα τα οποία θα παίξουν τον ίδιο ε, το, ρόλο ενός ε, σπόρου που θα μπορέσει να ε, αυξηθεί μετά, να μεγαλώσει, να παραγάγει. Εμείς θεωρούμε ότι το ΣΕΦ ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας είναι τουλάχιστον επί τρία για, τα, για τις χορηγήσεις και οχτώ για τα διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα, δάνεια κλπ και μπορούμε να φτάσουμε σε ένα, σε πολλαπλασιαστικό παράγοντα της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή μιλούμε εδώ για 20-25% του συνόλου των χρημάτων που θα χρειαστούν για την επένδυση στο ε, ευρύ φάσμα. Πολλά χρήματα, αλλά πολύ σημαντικά χρήματα. Δεν πρόκειται για χρήματα που θα διοικηθούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Το πρόγραμμα SEF ICT είναι έχει ως στόχο να αλλάξει την κοινωνία μας και για τα καλά. Έχει σχέση με την ικανότητα να προσφέρονται καλύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τις δημόσιες αρχές στους πολίτες, η δυνατότητα να διασυνδεθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την υποδομή cloud, το cloud computing δηλαδή, που αλλάζει πλέον τελείως τις βάσεις για, την, για τον ανταγωνισμό, για το cloud computing, δηλαδή η συνεργασία πολλών υπολογιστών, επιτρέπει στις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε πάρα, σε πάρα πολλά δίκτυα υπολογιστών. Οποιαδήποτε λοιπόν μικρά, μικρή ή μεσαία επιχείρηση, όπου και να είναι εγκατεστημένη, θα είναι το ίδιο ανταγωνιστική όπω οι μεγάλε επιχειρήσει. Και οι ΜΜΕ αυτέ είναι το ραχοκοκαλιά τη ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν είναι λοιπόν μόνο η υποδομή. Τώρα το ΣΕΦ αποτελείται από δύο στοιχεία. Τον τομέα τη υποδομή και τον τομέα των υπηρεσιών και αυτά έχουν σχεδιαστεί να πηγαίνουν χέρι-χέρι και πράγματι πηγαίνουν χέρι-χέρι. Δεν, υπάρχει, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν υπηρεσίε χωρί υποδομή και υποδομή χωρί την παροχή υπηρεσιών πάλι δεν έχει νόημα. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα λοιπόν των δύο πυλώνων αυτού του προγράμματο. Η πλευρά των υπηρεσιών έχει πανευρωπαϊκή διάσταση και αυτό το λέω διότι χωρί υποστήριξη από την Ένωση μου φαίνεται δύσκολο να προκύψουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες. Και εδώ μιλούμε ιδιαίτερα για πολίτες που κινούνται και, και επιχειρήσεις που κινούνται μέσα στο διαδίκτυο, όχι, όχι ε, σωματικά, όχι στην πραγματικότητα και να μπορούν να διακινούν τις παραγωγές τους μέσα στην Ευρώπη και να περνούν τις υπηρεσίες τους ψηφιακά από τη μια χώρα στην άλλη και η ε, δυνατότητα των πολιτών να μπορούν να κυκλοφορούν με τη λεγόμενη e-card, electronic card. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και βεβαίω όλα αυτά ξεπερνούν το απλό τεχνολογικό θέμα της ε, ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων. Αυτά τώρα βέβαια έχουν και ένα συγκεκριμένο ε, στόχο, δηλαδή η πανευρωπαϊκή διάσταση για τις ε, υπηρεσίες, ενώ η υποδομή έχει πολύ τοπικό χαρακτήρα και ιδίω η υποδομή που μιλούμε, όπου, μιλούμε, όπου μιλούμε για πρόσβαση. Η πρόσβαση στα δίκτυα είναι πολύ τοπική. Έτσι λοιπόν, ε, ναι, να έχουμε συνεργασία με έμπιστους εταίρους ε, τοπικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διασύνδεση, η πρόσβαση. Γνωρίζουμε ότι η συζήτηση σε FICT θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση για το δημοσιονομικό πλαίσιο, για το, τη χρηματοδότηση του MFF. Το FICT δεν είναι μονάχα δαπάνη χρημάτων, είναι επένδυση χρημάτων. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά έργα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν και θα υπάρξουν πολλά. Και στο τέλος θα θεωρηθεί επιτυχής η προσπάθεια αυτή. Για τις χώρες μέλη, ωστόσο, θα είναι χρηματοδοτικά ουδέτερη. Και σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, σκεφτείτε μονάχα τις εξοικονομήσεις που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και στον ιδιωτικό τομέα και στον κυβερνητικό τομέα και στον τομέα της υγείας ιδίως. Ε, εκεί οι εξοικονομίες στον τομέα της υγείας μπορούν να είναι σημαντικές. Δηλαδή να διατηρήσουμε το επίπεδο του κράτους πρόνοιας που διαθέτουμε σήμερα και να το βελτιώσουμε κιόλας για λιγότερα λεφτά. Εξετάζοντας το CFICT θα πρέπει να, εξετάσουμε, να το εξετάσουμε ιδίω υπό το φως του τι αποφέρει και τι ικανότητες έχει να επιτύχει εξοικονομήσεις του δημοσίου χρήματος. Θα τελειώσω λέγοντας τι θα γίνει εάν δεν προχωρήσει το CFRCT. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, 50 εκατομμύρια πολίτες μπορεί να μην έχουν βραχυπρόθεσμα ε, πρόσβαση στο ευρύ Και σύμφωνα με, τις, ε, με τους υπολογισμούς μας, ορισμένες εκατοντάδες θεσμών που λειτουργούν σήμερα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά έργα με την τεχνολογία cloud. Διακινδυνεύουμε μάλιστα μικρές και μεσές επιχειρήσεις να αποκοπούν από αυτή τη διαδικτύωση, αυτό το cloud technology. Και διαπιστώνουμε ήδη ότι δεν προχωρεί ταχαίως η Σχετικέ τεχνολογίες. Η Ευρώπη είχε πρωτοποριακό ρόλο στην εποχή της κινητής τηλεφωνία, του GSM. Τώρα αυτή η πρωτοπορία έχει χαθεί. Η πραγματικότητα αυτή είναι και οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και ενδιαφερόμαστε πολύ για το, για το έργο που ε, εκτελεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό και το παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ που μας δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ. Βόκτορα Βιόλα και ευχές για τη δουλειά σου. Συμπεράσματα ο συνάδελφος Κρότσμαν. Χωρίς μικρόφωνο. Ε, ε, Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτό που θα γίνει είναι για τη συνεργασία με τους συναδέλφους που θα έχουμε σίγουρα θα έχουμε ευκαιρία να συνεισφέρουμε πιο πολύ περαιτέρω για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Θέλουμε ένα τεχνικά, τεχνολογικά αναβαθμισμένο το δυνατόν περισσότερο επίπεδο για αυτά τα δίκτυα. Θα πρέπει να προσέξουμε, να μιλήσουμε να μην αποσυνδεθούν οι περιοχές της υπαίθρου. Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δίκτυα αποκινούμε τους συναδέλφους θα εκπονήσουμε συμβιβαστικές τροπολογίες για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε αυτούς τους στόχους και θα υποβάλουμε προτάσεις για χρηματοδότηση που πρέπει να συμφωνήσουμε επ' αυτών που θα διασφαλίζουν τη μέγιστη πρόσβαση σε αυτά τα ευρυζωνικά δίκτυα. Πρέπει να διασφαλιστούν κονδύλια για να επιτευχθούν όλα αυτά και πιστεύω ότι μπορούν να ε, ενστερνιστούν και να δεχθούν αυτές τις απόψεις οι συνάδελφοι και να προαχθούν αυτοί οι στόχοι. Χρειαζόμαστε αυτά τα ευρυζωνικά δίκτυα, τα ταχύτατα δίκτυα, διότι αυτά τα οποία γνωρίζουμε σήμερα ως δίκτυα, ήδη το 2020 θα είναι πλέον παροχημένα, θα έχουν ξεπεραστεί. Και θα πρέπει όλες οι χώρες οι οποίες εδώ καλούνται να δράσουν, να δούμε ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν. Η κυρία Τροτμαν είπε ότι δεν θα πρέπει να αγνοηθούν οι περιοχές της υπέθου. θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ταχύτερης, μεγαλύτερης ταχύτητας, ε, υψηλότερης ταχύτητας δίκτυα. Θα πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην εκπόνηση, στην πρόταση κάποιων συμβαστικών τροπολογιών. Δεν είναι τόσο δραματικό το θέμα, ούτε πρέπει να πάρει δραματικές διαστάσεις. Είναι δυνατό να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να επιτευχθεί αυτή η διασύνδεση των περιοχών της υπαίθρου με αυτά τα δίκτυα κάποιοι νέοι ορισμοί. Απορρίπτω μια τέτοια προσέγγιση. Θα επιβαρύνει και θα καταστήσει ακόμα πιο περίπλοκες και σύνθετες τις ε, διαδικασίες. Όλοι όσοι, αφορούν, ε, όσοι εμπλέκονται στην ε, εξέταση αυτών των θεμάτων έχουν απόψεις που θέλουν να συνεισφέρουν με αυτές. Ευχαριστώ λοιπόν όλους που συμμετείχαν και υποστήριξαν το έργο μου σε αυτό το εγχείρημα. Επιθυμούμε φυσικά όλοι να έχουμε μια ε, σημαντική και έντονη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αυτός είναι στόχος για μας που θέλουμε να επιτευχθεί και γι' αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε σε σχέση με δημόσιες για παράδειγμα ακροάσεις να μεριμνήσουμε ώστε να ακούσουμε τις απόψεις ε, των ιδιωτικών αυτών επιχειρήσεων, των κύκλων αυτών των επιχειρήσεων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρέπει να είμαστε ελαστικοί και ευέλικτοι και ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα διασφαλιστεί μια θετική συνεργασία. Ευχαριστώ για την ενεργό συμμετοχή και τις καλές προτάσεις των συναδέφων και των σκιωδών εισηγητών κυρίως. Ευχαριστώ. Τελείωσε η συζήτηση. Θυμίζω ότι θα ψηφίσουμε στις 5 Νοεμβρίου στην Επιτροπή και τον Ιανουάριο στην Ολομέλεια. Επόμενο σημείο αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2003-98 σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες σήμερα και το λόγο έχει ο συνάδελφος Κάλφιν που είναι εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να παρουσιάσω κάποια σύντομα στοιχεία που θα δείχνουν πού βρισκόμαστε επειδή ακόμα πρέπει να ε, καταλήξουμε στη γνωμοδότηση της Κοινοβουλικής Επιτροπής. Κάπου 130 τροπολογίες κατατέθηκαν και από ό,τι γνωρίζω σήμερα το πρωί μια αγγλική μετάφραση είναι διαθέσιμη. Ακόμα δεν έχει μεταφραστεί το κείμενο σε άλλες γλώσσες. Χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες για, για τα θέματα τροπολογιών μπορώ να σας δώσω την γενικότερη εντύπωση που αποκόμισα από τις προτάσεις των συναδέρφων και την γενικότερη στάση τους. Οι περισσότερες από αυτέ, θα έλεγα κατευθύνονται προς την γενική κατεύθυνση του να ανοίξουν οι πληροφορίες, να έχουμε ε, και εκεί που θέλει να πορευθεί η οδηγία αυτή την κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. Έχουμε όμως κάποια ευαίσθητα σημεία τα οποία έχουμε ήδη προαναφέρει και έχουμε εντοπίσει και θεωρούμε ότι δημιουργούν κάποιες ανησυχίες ακόμα και τη διαμόρφωση των τιμών, των τιμολογίων. Έχουμε κάποιες τροπολογίες που λένε τι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πακέτο για την πληροφόρηση και τις πληροφορίες και τα θέματα τιμολόγησης και για τις διεργασίες όσον αφορά την τεκμηρίωση και δικαιολόγηση των τιμών ε, θα πρέπει να υπάρξει λιγότερη επιβάρυνση, μικρότερη επιβάρυνση όσον αφορά την, τους παρόχους αυτών των πληροφοριών θα ήθελα να πάμε όμως λίγο πιο πέρα από αυτό το πλαίσιο. Αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε κάποια σημαντική αλλαγή με αυτή την οδηγία, θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια των κρατικών αρχών, των δημόσιων αρχών, να μην υπάρξουν υπερβολικές τιμές απρόσιτες τιμές και να μην καταχραστούν το ρόλο τους. Είναι πάλι εδώ το θέμα της ε, δημόσιας ε, ε, θέσης, κρατικής θέσης στις πληροφορίες και του ρόλου της. Και από την ομάδα μας και από τους σκιώδεις εισηγητές θα δούμε όλες τις τροπολογίες. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε συμβιβαστικές τροπολογίες με τον πιο ισορροπημένο τρόπο και πάλι θα πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα μπορεί να υποστηριχθεί συνενετικά από τους περισσότερους ε, από τα περισσότερα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Έχουμε τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν καταθέσει τροπολογίες. Η Επιτροπή Πολιτισμού έχει ήδη ψηφίσει επί των τροπολογιών της. Έχουμε και την ολοκλήρωση και ψήφιση στην Επιτροπή ίνκο και Νιούι. Κατά τα τέλη της εβδομάδας θα έχουμε όλες τις τροπολογίες και γνωμοδοτήσεις για την έκθεσή μας και θα τα δούμε όλα αυτά. Θα έχουμε και μεταφράσεις σε αντίτυπα ε, και που θα αρχίσουμε έτσι να, δούμε, να βλέπουμε τις, ε, τις συμβαστικές τροπολογίες. Το χρονοδιάγραμμα για την ε, εντολή, για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο θα εγκριθεί στις 5 Νοεμβρίου εδώ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή μας Ήτρε, στη συνεδρίασή μας που θα έχουμε τότε. Πιστεύω ότι μπορούμε να ετοιμαστούμε έγκαιρα και η πρόταση είναι να συνέθούν οι σκιώδεις εισηγητές πιθανότατα στο Στρασβούργο πρώτα για να δουν πρώτα τις τροπολογίες και τις δυνατότητες για συμβαστικές τροπολογίες ώστε να είμαστε έτοιμοι κατά τις αρχές Νοεμβρίου για να ψηφίσουμε τη δική μας γνωμοδότηση, τη θέση μας στην Ήτρε. Κατά τα άλλα, διαφορετικά έχουμε θέσει την πρώτη ημερομηνία κατά τα μέσα Νοεμβρίου για τον τριμερή διάλογο. 15η Νοεμβρίου θα είναι αυτή ημερομηνία. Τα καλά μαντάτα είναι ότι γίνεται η προσπάθεια να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και ή δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα και να κλείσει πριν από τα τέλη του έτους. Θα απαιτήσει αυτό πολύ ε, έντονη σε βάθος δουλειά. Αν είναι όμως πρόθυμο να προχωρήσει έτσι το Συμβούλιο είναι κάτι που πρέπει να εκτιμήσουμε και να προχωρήσουμε κι εμείς. Και πάλι λοιπόν, όπως είπα στο Στρασβούργο, θα ξαναδούμε το, τα, σχέδια των προτάσεων τροπολογιών. Στις 5 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Ήτρε για την εντολή για να περάσουμε στο τριμερή διάλογο. Στις 15 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, το χρονοπλαίσιο όπως προτείνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάλφιν. Ναι, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει προβλέψει και η Επίτροπη ή ο λόγος στους και όδης. Ο Σαλβατόρα Πρώτα, Επιθυμώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ. Κάλφιν για το έγγραφο που υπέβαλε. Όπως είπε, λάβαμε τις τροπολογίες μεταφρασμένες στα αγγλικά. Δεν είναι ακόμα η ώρα να στοχεύσουμε συγκεκριμένες τροπολογίες, αλλά νομίζω ότι σε συνεργασία με τον εισηγητή θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση στην Επιτροπή μας για τα βασικά θέματα σχετικά με τις χρεώσεις, τους ανεξάρτητους οργανισμούς και κάτι άλλο σημαντικό, σχετικά δηλαδή με τα αποκλειστικά δικαιώματα για, στην περίπτωση δηλαδή ε, ε, κοινοπραξίας δημοσίου ιδιωτικού τομέα για μουσεία και διάφορα αρχεία κλπ. Ο στόχος είναι να γίνει πιο διαθέσιμη η υπηρεσία αυτή, από πλευρά δημοσίων οργανισμών κυρίω, και γι' αυτό θα διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με το τι μπορεί να ε, χρηματοδοτηθεί. Οι τροπολογικέ δικέ μου έρχονται σε ένα από τα σημαντικά θέματα, να διευκρινίσουμε δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις θα υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτείται άνω του περιθωρίου του κόστους και ιδίω για τους δημόσιους οργανισμούς όπου ο νομοθέτης απαιτεί να αποφέρουν οι δραστηριότητες τους κέρδος. Και το ίδιο επίσης για συμφωνίες κοινοπραξιών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Καθώς επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε και την αναδρομική ισχύ της νομοθεσίας, ώστε να μπορέσει αυτή να καλύψει και κοινοπραξίες που ήδη λειτουργούν που ήδη ε, υπάρχουν. Θα συζητήσουμε συγκεκριμένα τις τροπολογίες και ελπίζω ότι οι σκιώδεις ηγητές και ο εισηγητής θα μπορέσουμε, δηλαδή στη συνεργασία μαζί τους, να καταλήξουμε όσο το δυνατόν συντομότερα σε συμβαστικές ε, τροπολογίες. Δεν βλέπω κανέναν από, την, από τους φιλελευθέρους. Για τους πρασίνους. Η Μάγια. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική εκπληκτική δουλειά του. Οι περισσότερες τροπολογίες από τους συναδέλφου είναι και αυτές πολύ καλές. Από μια αρχικά στεναρή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε τώρα πια την ευκαιρία να υποβάλουμε και εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο μια στεναρή δυνατή δική μας πρόθεση. Τούτων λεχθέντων έχω κάποια σχόλια. Στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων είπα ότι έκανε κάποια σχόλια το Συμβούλιο για την ε, τετρα, ε, τετράμινη περίοδο όσον αφορά τις διεργασίες αυτές. Ε, ενώ είναι ένα ανοιχτό πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δούμε πώς θα καθορίζεται ακριβώς το ανοιχτό πλαίσιο. Έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες που νομίζω ακριβώς ε, εκφράζουν τις ιδέες αυτές που θέλει να εκφράσει το Συμβούλιο, όμως δεν ε, αποκλείονται ανοιχτές δυνατότητες ε, πρόσβασης, open format και για να δούμε τι θα γίνεται σε σχέση με την διαμόρφωση των τιμολογίων ώστε να μην υπάρχει αντική επίπτωση. Σας ζητώ να υποστηρίξετε αυτές τις τροπολογίες που τροποποιούν τα άρθρα 2 και 5 5 αντίστοιχα και εκπλήσωμε πραγματικά για την απέτηση της τεχνολογικής ε, αμεροληψίας ή ουδετερότητας μέσα από τις τροπολογίες της ομάδας ΕΛΚΑ. Ουδετερότητα σημαίνει να μην διαφοροποιούμε μεταξύ ε, χάρτινης ε, ενημέρωσης και ηλεκτρονικής. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δουλεύουμε και με τις δύο δυνατότητες. Δεν είμαι αντίθετη, αλλά θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε υπέρ των ανοιχτών ε, διαστάσεων ή ανοιχτή πρόσβασης. Δεν είναι εύκολη η εφαρμογή όλων αυτών. Ο λόγος για τον οποίο εκφράζω αυτή την άποψη είναι ότι διαφορετικά μπορεί να επιβαρυνθούν και να αποβεί εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων που μπορεί να βρουν δυσκολίες ε, να είναι λειτουργικές σε σχέση με αυτές τις ε, προτάσεις. Σε σχέση με την προσιτή διαμόρφωση τιμών είναι κάτι σημαντικό. Δεν έχουμε καταθέσει επ' αυτού, ότι υποστηρίζουμε απόλυτα τον εισηγητή και την Επιτροπή σε αυτά τα σημεία. Επίσης με ικανοποίηση βλέπουμε ότι οι, από πλευρά των συντηρητικών ECR κατατέθηκαν τροπολογίες στην Ευνομική Επιτροπή για να διασφαλίζεται ότι από πλευρά του δημόσιου τομέα όταν υπάρχει τέτοια ψηφιοποίηση θα είναι δημόσια προσπελάσιμη όσον αφορά τους όρους που θα προβλέπονται ε, για την αποκλειστική χρήση μεταξύ ε, τέτοιων συμβασιούχων όταν θα λήγουν τέτοιου είδους συμβάσεις. Και αυτό το θέμα στην ε, Επιτροπή μας πρέπει να το δούμε. Θα ήταν αρνητικό εις δίτ οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να μην είχαν θετικές επιπτώσεις. Θέλω να επανέλθω στο θέμα των κρατικών εκπομπών οι κρατικοί πάροχοι υπηρεσιών εξαιρούνται από την οδηγία χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Ε, μπορούν με δημόσια κονδύλια να αποκομίζουν κέρδη. Και αυτό ε, ενώ έχει καλυφθεί η ε, δαπάνη εξακολουθούν και να θέλουν να σημειώνουν και ε, κέρδη. Ας υπάρξει μια ευκαιρία για νέους να συμμετάσχουν σε αυτά τα μέσα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κρατικό και που επί μεγάλο χρονικό διάστημα καθόριζαν την ανάπτυξη του δημόσιου κρατικού τομέα σε αυτές τις εκπομπές ε, κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Κάποιος που γεννήθηκε το 1945 ή πιο πριν γνωρίζει το τι συμβαίνει. Αυτό όμως δεν συμβαίνει για νεότερους όπως στην Ευρώπη για άλλους που είναι νεότεροι όπως εγώ που έχουν γεννηθεί μετά το, τη δεκαετία ας πούμε του 80 και σε σχέση με το ε, δασκλάινε κροκοντήλ που έχει προσαρτηθεί ακόμα και στη δική μου πατρίδα από ό,τι γνωρίζω για το 1980 το μόνο το οποίο να ε, έχει είναι η δυνατότητα αυτή ηλεκτρονικά να μπορεί να δράσει. Όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοιες κινήσεις ε, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα, το άνοιγμα της δυνατότητας πρόσβασης, πρέπει να δούμε αυτούς τους όρους. Όταν στη Σουηδία, για παράδειγμα, υπάρχει η προσπελασιμότητα online, ε, δεν μπορώ εγώ να την εκμεταλλευτώ και να χρησιμοποιήσω αυτή τη δυνατότητα, μια και βρίσκομαι στο Βέλγιο τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως θα μπορούσα να έχω πρόσβαση όταν θα επιστρέψω στη Σουηδία επιστρέφοντας μετά τη διαμονή μου εδώ. Όμως πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον για τους νέους Ευρωπαίους, να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο κοινή ταυτότητας που θα μπορέσει να απορρεύσει μέσα από αυτά τα ηλεκτρονικά ε, μέσα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και για τους κρατικούς παρόχους τέτοιου είδους εκπομπών. Είναι θέμα και κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Το χρειαζόμαστε έντονα. Δεν μπορείς ταυτόχρονα να ζητάς από τους νέους να μαθαίνουν την προηγούμενη ιστορία όταν τα πιο συνήθη θέματα για την πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες δεν είναι δυνατόν να είναι προσπελάσιμα και να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Να υποστηρίξουμε λοιπόν την ένταξη των δημόσιων παρόχων σε τέτοιες εκπομπές από πλευρά των κρατικών μέσων. Πολλά μπορούμε να κερδίσουμε, δεν θα χάσουμε τίποτα. Ευχαριστώ. Ε, δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις. Η Κομισιόν έχει Ευχαριστώ. Όπως και παλαιότερα, σε άλλες μου παρεμβάσεις, επιθυμώ να πω ότι η υποστήριξη που μας προσφέρει το Κοινοβούλιο μας ενθαρρύνει πολύ. Και ευχαριστώ ιδιαίτερο εν προκειμένου τον εισηγητή για την προθυμία του να προχωρήσει με την εργασία αυτή και να διασφαλίσει ορισμένες, ε, την σύνταξη ορισμένων συμβαστικών τροπολογιών ώστε να είναι έτοιμες για τον επικείμενο τριμερή διάλογο. Η ξεκάθαρη υποστήριξη του Κοινοβουλίου υπέρ των ιδεών που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν είναι ιδιαίτερα καλό δεχτή για μας και μας στηρίζει στις συζητήσεις που διεξάγουμε. Είναι γεγονός ότι λίγες χώρε μέλη δεν είναι ακόμα απόλυτα πεπισμένες σε ό,τι αφορά την αξία των ανοιχτών δεδομένων και σχετικά με τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει το άνοιγμα αυτό των δεδομένων για δημόσια χρήση. Πρόκειται λοιπόν για την τελική ευθεία που Πρέπει να διανύσει η ιδέα αυτή έτσι ώστε να γίνει δεκτή συνολικά και να λάβει νομοθετική μορφή. Είμαι ωστόσο βέβαιος ότι οι οι ευρωβουλευτέ που είναι παρόντε εδώ και παρούσε θα συνεργαστούν προ την κατεύθυνση αυτή. Ο συνάδελφος Κάλφιν θέλει και πάλι το λόγο για να ολοκληρώσει. Δύο λόγια μόνο, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά πραγματικά τους κοιόδης εισηγητές, ιδιαίτερα τον Σαλβαδόρ και την Αμέλεια, επειδή αυτό το θέμα το πήραν πολύ ζεστά και με όλη τους την καρδιά συμμετείχαν στις προσπάθειες. Αυτό πράγματι μπορεί να αλλάξει την, τα πλαίσια της δημόσιας επικοινωνίας και μπορεί να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για τους νέους. Τώρα, για το θέμα των δημόσιων εκπομπών, κρατικών εκπομπών, και παρόχων. Πρέπει αυτό την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που μόλις ακούσαμε να την πάρουμε ιδιαίτερα σοβαρά, διότι αυτό μπορεί να ανοίξει τεράστιες ευκαιρίες και πρέπει φυσικά να δούμε αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να, να αντιμετωπιστούν τα θέματα και πνευματική ιδιοκτησία σχετικά, αλλά όσο πιο προσπελάσιμη και πιο προσβάσιμη είναι αυτή, αυτού του είδου η πληροφόρηση, τόσο πιο θετικό θα είναι αυτό. Και πάλι πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να προτείνουμε κάτι να προτείνουμε κάποιους συμβιβασμούς, συμβαστικές τροπολογίες που δεν θα αποδυναμώσουν, δεν θα νερώσουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα δημιουργήσουν ένα στεναρό, ένα δυνατό πλαίσιο ως θέση που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε με αυτό το σημείο. 5 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε. Τελειώνουμε τις εργασίες μας για σήμερα το πρωί. Θα ξεκινήσουμε τις ε, τρεις ε, σήμερα το απόγευμα σχετικά με την ε, κυρία Γιογκέχαν Κουίν, την Επίτροπο για την Έρευνα και την Κοινοτομία, σχετικά με την έρευνα.